Good morning, Καλημέρα σας. Να επαναλάβουμε τις εργασίες μας σήμερα. Έχουμε το μέλλον των καθεστώτων ελέγχου των πυρηνικών όπλων και τις επιπτώσεις για την ασφάλεια της Ένωσης ως επόμενο θέμα στη Μερσιά Διάταξη. Είχαμε μια πρόσφατη ανταλλαγή από με την καμίτσου, Ιζούμι Νακαμίτσου, αναπληρώτρια γενική γραμματέα και πάτε εκπρόσωπο ε, για τα θέματα εξοπλισμού σε επίπεδο ΟΗΕ για τις ε, προοπτικές ε, της διάσκεψης εξέτασης αυτής της ε, συνεχιστικής διάδοση του 2027 με 22 Απριλίου με 22 Μαΐου στη Νέα Υόρκη. Αυτή η συνθήκη είναι ακρογωνίως λίθος της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για τη μη διάδοση και τον πυρηνικό αποκλεισμό. Είναι το μόνο δυναμικά δεσμευτικό μέσο με βάση τη συνθήκη υπέρ της, ε, του πυρηνικού αφοπλισμού, της ασφάλειας σταθερότητας, αλλά για να πετύχει το βασικό στόχο πρέπει να πετύχει κάποιου ενδιάμεσου στόχο. Είναι μια βαθμιδόν προσέγγιση, το step by step ε, που είναι ο βασικός ε, πυλώνας της συνθήκης που δέχτηκαν τα συμβαλόμενα μέρη το 70 όταν και τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη Υπάρχει το ΤΑΙΣ που είναι η συνθήκη πλήρους απαγόρευσης των πυρνικών δοκιμών, ένα σημαντικό στάδιο. Δεν έχει ακόμη όμως τεθεί σε ισχύ 184 χώρες έχουν υπογράψει, 168 έχουν επικυρώσει και τρία κράτη εξ αυτών έχουν πυρηνικά όπλα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο. Για να τεθεί σε ισχύ θα πρέπει ακόμη να επικοινωθεί από 8 χώρες, Σε Ινδία, Πακιστάν, Κίνα, Αίγυπτο, Σιράν, Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε στήριξε ε, και απίφθηνε έκκληση για την κύρωση στις χώρες που δεν το έχουν κάνει. Παραλληλώς έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες να προωθήσουμε μια γρήγορη ε, σύναψη συμφωνίας για τα σχάσιμα υλικά. Διεθνή συμφωνία που απαγορεύει την παραγωγή ουρανίου και εμπλουτισμένου πλουτονίου. Επιβάλλονται νέες, ε, επίσης, νέοι περιορισμοί στη ΣΥΠΑ, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κίνα που έχουν ε, πυρηνικά όπλα και η Ισραήλ, η Ινδία, Πακιστάν και Βόρεια Κορέα, τέσσερα κράτη που έχουν πυρηνικά όπλα αλλά δεν έχουν υπογράψει τη συμβεστιμή διάδοση. Σε διεθνές ε, επίπεδο τώρα, ε, λόγω της αβεβαιότητας και που έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν την πυρηνική απειλή ως μοχλό για αποσταθεροποίηση και εκβιασμό, όταν έχουμε κράτη σημαντικά τα οποία παναχωρούν από τις δεσμεύσεις, απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια ισορροπία, στην επόμενη διάσκεψη εξέταση της ε, ε θα πρέπει να δεσμευτούν τα κράτη με βάση συγκεκριμένε προτάσεις για να προωθήσουν ε, τη μη χρήση πυρηνικών όπλων ως απαραβία στο δεσμευτικό κανόν και να λάβουν υπόψη τους την κατάσταση ε, που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά σε χρήση του πυρηνικού όπλου και βέβαια αυτό θα ε, θέσει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο τη στρατηγική ισορροπία σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν δύο διμερεί σημαντικά μέσα ε, ΗΠΑ Ρωσίας ε, για τη σταθερότητα και τη στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών, το INF και το New Start. Είπα ανακοίνωσαν ότι αποχωρήσουν από ε, την ε, συνθήκη ε, για τις πυρηνικές δυνάμεις το Φεβρουάριο του 19. Εμείς ζητούμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλωμένων για να σωθεί ε, αυτή η συνθήκη, το INF δηλαδή, και θα γίνουν συστάσεις για τη διάσκεψη που θα ε, ψηφιστούν αύριο στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Επίσης έχουμε το New Start. Ε, παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση μια ακόμα δημερού συμφωνίας. Θεωρούμε ότι θα ήταν καλό ε, να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ακρόασή μας θα συνοδεύεται από μια ανταλλαγή απόψεων για δύο θέματα που κυριαρχούν στη συζήτηση και που είναι και θέματα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα και τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για το Ιράν και τις υποχρεώσεις της Τεχεράνης και κατά δεύτερον τις πρόσφατες πυρηνικές δραστηριότητες της ε, Κορέας. Πώς θα οργανωθεί η ακρόασή μας. Καταρχάς θα έχει το λόγο κυρία Άντζελα Κέιν, που είναι υπεύθυνη για την έρευνα ε, στη Βιέννη, ε, στο κέντρο για τον αφοπισμό και τη μη διάδοση. Έχει διατελέσει και είπατε πρόσωπος ε, για τα θέματα αφοπλισμού στα Ηνωμένα Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε την διάσκεψη εξέταση της συνθήκης του 2020 και πώς θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα το μέλλον σε ό,τι αφορά τον κόσμο έλεγχο των πυρηνικών 10-15 λεπτά σας φτάνουν. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την ε, συνεδρίαση, σε αυτό το φόρουμ. Θα μιλήσω αγγλικά. Θέλω να θέσω το πλαίσιο γιατί νομίζω είναι σημαντικό να υπενθυμίσω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Μιλήσατε για την κατάργηση της συμφωνίας για τα όπλα, την ε, συνθήκη δηλαδή μη διάδοση των πυρηνικών. Επίσης, είχαμε την ε, διείσδυση στην ε, Κορέα, πολιτικές ε, ανακατατάξεις, ε, ένταση στη Μέση Ανατολή, ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις στον στρατιωτικό εξοπλισμό και την τεχνολογία και στα πυρηνικά και έχουμε όλο και μεγαλύτερους κινδύνους λόγω των πιθανών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης, έχουμε μια κατάσταση όπου αυτά που ήταν δεδομένα κάποτε σε ό,τι αφορά τις ε, συμμαχίες και τα πολυμερή συστήματα δεν ισχύουν πια. Να σας ε, δώσω κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα, πολλοί από σας τα ξέρετε. 75% ε, αυξήθηκαν οι δαπάνες για τα στρατιωτικά τα τελευταία 20 χρόνια. 75%. Είμαστε στο 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι μια αύξηση 2,6% σε σχέση με το 2017. 2,6% δεν είναι πολύ, δεν μοιάζει πολύ. Αλλά αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για 1,8 τρισεκατομμύρια, είναι τεράστιο. Και οι πέντε δυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ε, Κίνα, ε, Σαουδική Αραβία, Γαλλία. Ε, στον ε, προϋπολογισμό του 2021 των Αμερικανών, οι Αμερικανοί μας είπαν ότι θέλουν να έχουν... Ε, αύξηση 19%, ε, 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ε, αύξηση πάνω από 50% σε σχέση με το 2017, ε, που ήταν η πρώτη χρονιά του Τραμπ στην εξουσία, με νέα υποβρύχια εκτόξευσης πυρηνικών κεφαλών. Θέλουν να συγχρονίσουν τα συστήματα εκτόξευσης πυρηνικών. δεν έχουμε πλέον την συμφωνία μη διάδοσης και δεν έχουμε και άλλες διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία εκτός από το New Start. Όταν κοιτάξτε το ε, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που έχει την περασμένο μήνα, βλέπετε τα τελευταία τρία χρόνια ε, τα όπλα μαζικής καταστροφής ήταν πάνω-πάνω στην ε, λίστα και όμως το Οικονομικό Παγκόσμιο Φόρουμ, λόγω της οικονομικής εστίασής του, δεν θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα και για τις επιπτώσεις του θέματος. Τον Ιανουάριο ε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει πιο, από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε φτάσει πιο κοντά στην ημέρα της αποκάλυψης. Κάθε πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ε, Κέννεντι κάνει συνθήκες με την ε, Σοβιετική Ένωση ή με τη Ρωσία και όμως δεν περιορίζονται πυρηνικέ δοκιμές, που, κάτι που ανέφερε και η Πρόεδρος. Ε, οι Ευρωπαίοι είχαν, υποστήριζαν τη συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών πολύ έντονα. Παρά όλα αυτά, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Ε, υπάρχει ένα στρατηγικός ανταγωνισμός χωρίς πόλεμο. Ε, οι συμφωνίες αυτές ή η απουσία συμφωνιών δεν γίνεται μέσα σε ένα κενό. Ε, αυτοί που επιβλέπουν την παραγωγή όπλων ε, ανακοίνωσε ότι ε, έχουμε παραγωγή πυρηνικών ε, πιο αδύναμο, κατά το 1 τρίτο, ε, σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη Χειροσύμα που θα μπορούσε να είναι έτοιμο ε, προς ανάπτυξη εντός μηνών. Αν το συνδυάσουμε με την αναθεώρηση του 2018 για τα πυρηνικά των Αμερικανών, άλλαξαν τον ορισμό για αυτό που λένε ακραίες συνθήκες, ε, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε θα χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά όπλα, όπως μη πυρηνικέ στρατηγικέ επιθέσεις ή πυρηνικέ επιθέσει εναντίον μιας ομάδας, όπως λένε, που υποστηρίζουν τις, σε περίπτωση μάλλον που έχουμε τρομοκρατικέ απόπειρε για απόκτηση πυρηνικών. Ε, επίσης, ε, θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικά όπλα σε περίπτωση μη πυρηνικών ε, στρατηγικών υποθέσεων εναντίον των ΙΠΑ ε, ή εναντίον της υποδομής του πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την ε, περίπτωση χρήσης ε, πυρηνικών στο παρελθόν. Ε, μετά την αναθεώρηση της ε, χρήσης των πυρηνικών από τις ΕΠΑ και ο Πούτιν το Μάρτιο του 2018 ανακοίνωσε υπερηχητικό πύραυλο, την κατασκευή υπερηχητικού πυράβλου, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι η κατάσταση ακόμα, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες σχέση με αυτό. Δεν έχω χρόνο. Προσπαθώ να πω όσο περισσότερα μπορώ. Now, um, Μετά την κατάργηση ε, της ε, συνθήκης για τη μη διάδοση, ε, έχουμε το New Start, όπως είπε και η πρόεδρος, που είναι η μόνη συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών μεταξύ Αμερικανών και Ρωσίας και εκπνέει το Φεβρουάριο του 2020, ένα μήνα μετά την έναρξη της ε, νέας ε, προεκλογικής εκστρατείας για τον νέο πρόεδρο. Τέλη του 19 είχαν ξεκινήσει οι προϋποθέσεις για την παράταση του New Start για πέντε χρόνια. Ε, οι Αμερικανοί δεν έχουν ανταποκριθεί όμως και ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα ήθελε να ονομάσει ένα διαπραγματευτή ψηλού επίπεδου για να επιβλέψει τι ε, πυρηνικέ συνομιλίε με την ε, Ρωσία και πιθανώ με την Κίνα. Πού βρίσκεται η Ευρώπη τώρα. Όπως ξέρουμε, η συνθήκη για τη μη διάδοση ε, ε εξάλληψε μία ολόκληρη κατηγορία όπλων, αλλά δεν υπήρχαν διαβουλεύσεις με την Ευρώπη. Η κατάργηση της, μιας άλλης συνθήκης για τα πυρηνικά άφησε τους Ευρωπαίους ε, σε μια αναζήτηση για την μετέπειτα κατάσταση. Μιλάμε για την απαγόρευση, μάλλον μιλάμε για την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. με τι έχουμε να κάνουμε λοιπόν τώρα. Τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής Αμερικανός υπεύθυνο για τα πυρηνικά και, την, και τον αφοπλισμό, Chris Ford, ε, μίλησε πάρα πολύ έντονα και πολύ εχθρικά για το πού ε, βρίσκεται η Αμερική σε σχέση με τη συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών. Πολύ εχθρική γλώσσα, ειδικά προς τους υπερασπιστές ε, και οι θειασότες της συνθήκης μη διάδοσης. Για όσους θέλουν αυτή τη συνθήκη NPT, δηλαδή τη συνθήκη μη διάδοσης, να γιατί είναι το μόνο εργαλείο που εμποδίζει τη διάδοση. Η φρασιολογία που χρησιμοποιείται, που είναι εχθρική μπορώ να το πω, εναντίον αυτών που δεν συμφωνούν με τους πυρηνικούς στόχους των Αμερικανών, καθιστούν πολύ δύσκολο ε, το έργο της εξέβρεσης συμφωνίας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που είδα ότι είναι πολύ θετικές. Ε, ε μια ομάδα ανάπτυξης ε, πυράβλων που ξεκίνησε ως ε, ε, προσπάθεια από τη Γερμανία, νομίζω, και είναι χρήσιμη πρωτοβουλία. Η πρόεδρος ανέφερε την συνθήκη για την απαγόρευση του, του σχάσιμου υλικού. Είναι πάρα πολύ σημαντική συνθήκη και υπάρχει και η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην επαλήθευση των πυρηνικών ε, στα θέματα διαφάνειας. Θα βοηθούσε πάρα πολύ, όχι μόνο για την Ευρώπη, ε, αλλά και τα κράτη-μέλη της ε, συνθήκης που έχουν υπογράψει, τα, τα κράτη-μέλη της με διάδοση των πυρηνικών. Θα μπορούσε να αλλάξει τους στόχους παρά να περνάμε σε αντεγκλήσεις και να μιλάμε συνέχεια για περιβάλλον αφοπλισμού, γιατί κανένας δεν ξέρει αν έχουμε κάνει αν έχει νόημα να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στο παρελθόν, α πούμε, είχαμε κάνει όλα τα βήματα, είχαμε τι προποθέσει ε, για τον αφοπλισμό και τελικά τίποτα δεν έγινε. Επίση, χρήσιμο θα ήταν να ξεκινήσει διάλογο με τη Ρωσία, κατά την άποψή μου, γιατί όπω ξέρουμε, ήταν κατά τη ε, μονομερού ε, κατάργηση τη συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών και θα πρέπει να δούμε και τι επιπτώσει από την κατάργηση τη Συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών τη NPT. Πού βρίσκεται η Ευρώπη, πώ θα την επηρεάσει αυτό την Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να, συμβουλευτούν, να διαβουλευτούν με τους συμμάχους, αλλά αν υπάρχει ανάπτυξη πυρηνικών θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους Ευρωπαίους κυρίως εταίρους. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το ΝΑΤΟ. Ε, γιατί μερικέ φορέ υπάρχουν και επικαλύψει ανάμεσα στο ανήκει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Επίση, το ΝΑΤΟ έχει πυρηνικά όπλα εδώ στο Βέλγιο και σε άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Και είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το οποίο θα πρέπει να τεθεί. Το ΝΑΤΟ ως συμφωνία, συμμαχία, ε, αποφάσισε ότι θα παραμείνει πυρηνική όσο υπάρχουν πυρηνικά, ε, είναι μια πολύ έντονη δήλωση που έχουν προσυπογράψει οι συμμετέχοντες στο ΝΑΤΟ. Ε, επίσης, ε, μέχρι το 2024 θα πρέπει να αλλάξουν τα αεροπλάνα που φέρουν πυρηνικά όπλα ε, του ΝΑΤΟ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, με τις εκτοξεύσεις, θα γίνει ε, και οικονομικά με αυτό το θέμα, αυτή την αλλαγή. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ευρύτερο διάλογο για τη στρατηγική σταθερότητα. Όλοι κοιτάνε τα πυρηνικά, λες και είναι τα φοβερά όπλα, αλλά με τις νέες τεχνολογίες, με τους υπερηχητικούς πυράβλους και με άλλα όπλα, νομίζω ότι υπάρχει ένα ποιοτικό άλμα στις δυνατότητε ανάπτυξης ε, όπλων. Και κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς αυτό θα επηρεάσει τα πράγματα ε, και πώς θα επηρεαστεί η στρατηγική σταθερότητα από αυτό. Έγινε μια προσπάθεια πέρυσι στα τέλη από το Βέλγιο και του χρόνου και τη Γερμανία, ε, δύο χώρες που έχουν πυρηνικά και συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και είναι και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να υπάρξει ένας διάλογος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όχι γιατί θα ξανακούσουμε τις ίδιες θέσεις που έχουμε ξανακούσει, αλλά γιατί και άλλα κράτη-μέλη θα έχουν έτσι την ευκαιρία να πούν τις απόψεις τους και νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί οι συζητήσεις μέχρι στιγμής περιορίστηκαν. Ε, όλοι ακούμε τα ίδια και τα ίδια σαν ηχό ας πούμε. Και πέρυσι ε, το ζήτησε η Κίνα και η Ρωσία, περίεργος πώς, μία συνάντηση στο ΝΟΙΕ για τους ε, πυράβλους κρούς μεσαίου βεληνικούς ε, και, και τις δοκιμές που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. επαναλήφθηκαν οι, οι διαστάσεις, αλλά το βασικό είναι να ακουστούν και νέες απόψεις οι οποίε ακούστηκαν επίση. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μέτρα μείωση του κινδύνου. Ε, η προσπάθεια που έγινε δυστυχώ μετά το 2010 για την, με βάση την πρωτοβουλία της Νορβηγίας για, την, για τις συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης, ε, παρότι είχαν γίνει πάρα πολλά, ε, μπήκαν λίγο στο περιθώριο. Καλό είναι να βιώσει λιγάκι αυτή η προσπάθεια, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται αν εκραγούν ας πούμε, τα πυρηνικά σήμερα, μια κατάσταση που είναι τελείω διαφορετική από αυτή που θα είχαμε πριν από 10 χρόνια. Μια άλλη σημαντική συνεδρίαση έγινε πέρυσι τον Ιούνιο σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Ε, την ε, οργάνωσε η Σουηδία ε, και συμμετείχαν και χώρε που δεν έχουν πυρηνικά και ασχολήθηκε με τη συνθήκη με διάδοση των πυρηνικών. Τι μπορεί να γίνει ε, για την NPT, για αυτή τη συνθήκη με διάδοση των πυρηνικών ζωφερή κατάσταση. Όλοι λέγανε τι σημαίνει αυτό, μιλούσαν για ένα έγγραφο συνένεση, υπάρχει τελικό κείμενο, δεν έχουμε τελικό κείμενο, λέγανε όλοι. Και αν όχι, ε, και αν για δεύτερη φορά δεν υπάρξει ε, πάλι έγγραφο, τι θα γίνει και τι σημαίνει αυτό την πεντηκοστή επέτειο από τη θέση ισχύ της NPT. Ε, υπήρχε μια δυνατότητα συντονισμού της θέσης εντός της Ευρώπης ε, και όταν τη λέω Ευρώπη, ε, φυσικά δεν μιλάω για ε, χώρες που έχουν πυρηνικά, αλλά και για μέλη του ΝΑΤΟ και για χώρες που δεν έχουν πυρηνικά και που απαγορεύουν τα πυρηνικά. Αυστρία, Ιρλανδία π.χ. Θα ήθελα να αναφέρω και μια τελευταία προσπάθεια, η δημόσια στήριξη για τον αφοπλισμό. Πρόσφατα έγινε μια δημοσκόπηση του κοινού και πάνω από το 80% των νέων είναι αντίθετη με τους, με τους πυρηνικούς εξοπλισμούς. Πάνω από 80% εντυπωσιακό μου φαίνεται που είναι τόσο ψηλό αυτό το νούμερο. Ε, και το βλέπουμε και τη σύγκληση που υπάρχει ανάμεσα στον, στον έλεγχο το, των όπλων και του αφοπλισμού και το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον ε, έχει, υφίσταται πάρα πολλές συνέπειες λόγω των πυρηνικών και τη συγκέντρωση των πυρηνικών. Αυτά θα σταματήσω εδώ και αν έχετε ερωτήσει να επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πλουσιότατη παρουσίαση. Ο Μάρκ Φίλιπς είναι εμπειρογνώμων σε θέματα ε, πυρηνικών. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται με τον ε, αφοπλισμό σε διατλαντικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τη συνθήκη μη διάδοσης ε, διότι αυτή τη στιγμή το μέλλον της είναι αβέβαιο ε, και είναι πολύ σημαντικά τα πράγματα αυτά. Να σας δώσω αμέσω το λόγο. Καλημέρα. Θα μιλήσω για ένα στοιχείο στο καθεστώς της συνθήκης μη διάδοσης, το οποίο είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Η συζήτηση γίνεται κυρίως στη Βιέννη, όχι εδώ στις Βρυξέλλες. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία γι' αυτό, μπορεί και να τα γνωρίζετε κάποια από αυτά. Αν όντω τα γνωρίζετε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων και μετά θα κάνω κάποια σχόλια για το ρόλο των Ευρωπαίων ε, σε αυτή τη δύσκολη ε, απόφαση. Στις 9 ε, Μαρτίου, ο νέος διευθυντής Μάρκο Γκρόση της Επιτροπής για τον ε, ζήτησε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν η τελευταία συνάντηση για να δούμε την κατάσταση στο Ιράν. Και η συνθήκη μη διάδοση είναι αυτή η οποία θα δώσει το πλαίσιο για τη συζήτηση αυτή. Όπω γνωρίζουν κάποιοι από εσά, πριν από ένα ακριβώ χρόνο, το Ιράν ε, φιλοξένησε μία συμπληρωματική επίσκεψη στην οποία έδωσε πρόσβαση σε πυρηνικέ εγκαταστάσει. Ε, και η ε, Διεθνής ε, ε, Ατομική Υπηρεσία πήρε και κάποια δείγματα και είδαν ότι υπήρχαν σωμα επεξεργασμένου ουρανίου που φαίνεται ότι ήταν διαδικασίες εμπλουτισμού ουρανίου και μετατροπής ουρανίου. και οι περιοχές αυτές δεν είχαν δοθεί δημοσίως και μέχρι τώρα οι προσπάθειες της υπηρεσίας, της Διεθνούς Ατομικής Υπηρεσίας να λάβει στοιχεία για τα θέματα αυτά που το Ιράν δεν έχει αποφέρει καρπούς. Θα πρέπει να δοθούν αυτές οι πληροφορίες ώστε να επιβεβαιωθεί εάν ε, τα πορίσματά της ε, υποδεικνύουν ότι υπάρχει υλικό ε, στο Ιράν και δεν έχει υπάρξει συνεργασία με την υπηρεσία από πλευρά Ιράν. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να το επιτύχουν. Αυτή είναι η υποχρέωση του Ιράν βάσει τη ε, Συμφωνία Μη Διάδοση ε, Όπλων. Ε, το Ιράν συμμετέχει στη συνθήκη από το 1994 και αυτό διευκρινίζεται στην παράγραφο 7 τη Συμφωνία για τι Δικλείδε Ασφαλεία τη Συμφωνία Μη Διάδοση. Στο παρελθόν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα κράτη-μέλη της Υπηρεσίας ε, έχουν ε, ε, συμφωνήσει ότι πρέπει να δίνονται αυτές οι πληροφορίες όταν τη ζητά η υπηρεσία. Όλα αυτά εκτιλήσονται σε μια στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικαλεστεί το DIM για την συμφωνία. Το Ιράν απειλεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία αν αποφασιστεί να παραπευθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό που έχει σημασία για την όλη συζήτηση και πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το θέμα αυτό το οποίο αντιμετωπίζει το Δικητικό Συμβούλιο στη Βιέννη αυτή τη στιγμή δεν αφορά τις δεσμεύσεις του Ιράν για τη συμφωνία, αλλά τη συμφωνία μη διάδοση όπλων και δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγχυση μεταξύ τη συμφωνία με το Ιράν και τη συμφωνία μη διάδοση όπλων η συμμόρφωση με τις δικλείδες ασφαλείας είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου των ε, κρατών μελών. Βάσει λοιπόν των διαδικασιών, σε μια τέτοια περίπτωση, αν το Δικαιωτικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι μια χώρα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της, η συνήθις διαδικασία είναι το θέμα αυτό να παραπευθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και δεν υπάρχει κάποια ε, εικόνα για το κατά πόσο θα συμβεί. Δεν είναι σαφέ αν θα συμβεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κομβικό ρόλο σε αυτό το σημείο. 35 κράτη-μέλη της Υπηρεσίας ε, ε, Ατομικής Ενέργειας ε, ε, είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν και τα 17 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρέσβης της Σουηδίας ε, στην υπηρεσία είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 7 Δεκεμβρίου ε, έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση της υπηρεσίας για να συζητήσει το θέμα, διότι δεν μπόρεσε να λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεται από το Ιράν. Και υπήρξαν δηλώσεις από τα κράτη-μέλη ε, τα οποία ήταν αναφανδόν υπέρ της τάσης της γραμματείας επί του θέματος αυτού. Ήταν αντίθετη ε, μόνο κάποιες δηλώσεις ε, της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι οποίες για δύο λόγους είχαν αποκλίνουσες απόψεις. Η μία είναι ότι οι Ρώσοι δήλωσαν στη γνωμοδότησή τους ότι το εν λόγω υλικό στο Ιράν παρήχθη από το Ιράν πριν από δεκαετίες και επομένω δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει σχέση με τη σημερινή συζήτηση και επίσης ε, είπαν ότι η υπηρεσία ατομικής ενέργειας ε, εάν λάβει μια μεσοπρόθεσμη απόφαση ε, για το θέμα αυτό, θα αποτελεί διάκριση για κράτος μέλος της υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αυτής της άποψης Και εδώ θα ήθελα να τονίσω για τους σκοπούς αυτής της συζήτησης ότι το σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο συζητούμε αυτή την εβδομάδα, περιλαμβάνει κάποια σημεία τα οποία έχουν άμεση σχέση με το θέμα αυτό. Αν δείτε το σημείο 1α, γίνεται μία ε, στη διεθνή τάξη βάση κανόνων. Είναι προϋπόθεση για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Πολλοί από εσά μπορεί και να γνωρίζετε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία σε αρκετές περιπτώσεις ε, και μάλιστα πρόσφατα έχει δηλώσει ότι αυτή η διεθνή τάξη βάση κανόνων είναι μια δυτική επινόηση για να κάνει διακρίσεις κατά κρατών και να υποχρεώνει κράτη να κάνουν πράγματα τα οποία δεν υποχρεώνται στην πράξη να κάνουν και μέσω των υποχρεώσεών τους ε, στην υπηρεσία ατομικής ενέργειας η Γραμματεία της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκφράσει την άποψη ότι ο, η υπηρεσία υποχρεούται βάσει της συμφωνίας για τις δικλείδες ασφαλείας του Ιράν και μετά όσων έχουν ε, ψηφιστεί σε προηγούμενα ψηφίσματα να προχωρήσει το θέμα ε, του Ιράν. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο περιλαμβάνεται στο σχέδιο σύσταση και έχει άμεση σχέση και σε μεγάλο βαθμό μετά τα όσα συζητούμε. Αν δείτε το σημείο 1K έως 1N, εκεί θα δείτε ότι υπάρχει αναφορά ώστε να πιεστούν οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε και η, η Ρωσία να αναλάβουν ευθύνε κυρίω όσον αφορά τα πυρηνικά ζητήματα, όπω πολύ σωστά επεσήμανε η Άντζελα. Και αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο στη Βιέλη αποκαλύπτει ότι οι Ηνωμένε και η Ρωσία πρέπει να ε, θυμηθούν τι υποθέτει η Συμφωνία για τη μη διάδοση και τη τήρηση των δικλείδων ασφαλείας και εάν δεν υπάρχει συνεννόηση για το ε, ποιο είναι το σημείο από το οποίο μια χώρα θα θεωρείται ότι είναι απειλή για πυρηνική διάδοση στο παρελθόν, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και ε, στη συνέχεια, υπήρχε μια τέτοια συνεννόηση μεταξύ Πολιτείων και Ρωσία. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και πρέπει να προειδοποιήσουμε και τι Πολιτείε και τη Ρωσία ότι είναι αυτό απαραίτητο. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ένδειξη ότι το σύστημα έχει διαραγεί. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ε, μια μεσοπρόθεσμη απειλή διάδοση. Η Ρωσία θεωρεί ότι δεν είναι απειλή μεσοπρόθεσμα. Γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι το σχέδιο σύστασης το οποίο έχετε ενώπιόν σας θα πρέπει να τροποποιηθεί για να πάει πέρα του θέματος της, του αφοπλισμού από τα πυρηνικά όπλα και να περιλαμβάνει και τη μη διάδοση και τις δικλείδες ασφαλείας ως ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προσέξουν αυτοί που θα συμμετέχουν στη διάσκεψη αναθεώρησης της Συμφωνίας Μη Διάδοσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όπως λέει το σημείο 1ΑΑ στη σύστασή σας και παραθέτω, επιβεβαιώνω τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε εξασφαλίσει για ε, ειρηνικό και η χρήση πυρηνικών ε, από το Ιράν και να υπενθυμίσουμε στο Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στις συμφωνίες και τη συμφωνία με διάδοση πυρηνικών. Θα πρέπει να υπάρχει τέτοια διατύπωση σε αυτή τη σύσταση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Συμφωνία Μη Διάδοσης και οι υποχρεώσεις του Ιράν βάσει της Συμφωνίας Μη Διάδοσης που εκφράζεται στη Συμφωνία για τις Δικλείδες Ασφαλείας είναι η βάση για τη συμφωνία ε, με το Ιράν. Δεν είναι ξεχωριστά πράγματα και θα είναι και αυτό το οποίο θα περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία κάνει το Ιράν με άλλα ε, κράτη για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και στην Ευρώπη για τη δημόσια συζήτηση από αυτού, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, κυριαρχείται από την ε, ανησυχία για την διάσωση της συμφωνίας με το Ιράν για την ασφάλεια της Ευρώπης, αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να υπάρχει επαλήθευση και να ε, υπάρχει και η συμφωνία για τις δικλείδες ασφαλείας και να δούμε και τι γίνεται με τη συμφωνία με το Ιράν. Τέλος, να πω εδώ στην εισαγωγή μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια πηγή πληροφοριών για τη μη διάδοση έχει μεγάλη εμπειρία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτές τις πληροφορίες να τις θέσει επιτάπητος στη συζήτηση και με τις πολιτείες και με τη Ρωσία προκειμένου να υπάρξει αυτή η κοινή συνεννόηση όπως σας είπα. Πώς θα γίνει αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επαφίεται στα μέλη της ηθίκης και θα πρέπει να τα αποφασίσουν αυτοί. Αλλά θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε εδώ ότι πολύ συχνά, όπω γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 να καταλήξει σε κοινή θέση για το τι θεωρείται ο τρίτη ε, πυλώνα της συμφωνίε μη διάδοση, δηλαδή την ειρηνική χρήση τη πυρηνική ενέργειας. Αυτό είναι πρόβλημα και πρόκληση για εσά, γιατί υπάρχουν ε, χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν με επιτυχία πυρηνική ενέργεια και άλλε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμμερίζονται την άποψη ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ασφαλής και βιώσιμη. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε θέσεις οι οποίες να έχουν στρατηγικό αντίκτυπο επί του θέματος. Θα ήθελα εδώ να σκεφτείτε και το εξή. Στην περίπτωση που σας παρουσιάζω εδώ σήμερα, δεν τίθεται τέτοιο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 συμφωνεί από αυτού. Είμαι 100% βέβαιος. Η θέση που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέφρασε το Νοέμβριο για στήριξη της γραμματείας είναι συνενετική θέση. Δεν υπήρξαν φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, είχα, να έχουν διαφορετική άποψη από τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 27. Επομένως είναι κάτι από το οποίο συμφωνείτε όλοι, είστε ενωμένοι από αυτού και σας προτρέπω να χρησιμοποιήσετε αυτό το γεγονός για να προχωρήσετε στις συζητήσεις σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Ρωσία ώστε να πιεστούν να ε, συμμετέχουν και να δεσμευτούν για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλάρα Πορτέλα. Για πείτε μας εσείς πώς βλέπετε το μέλλον του έλεγχου των πυρνικών όπλων και πώς ε, θα επηρεάσει μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα την Ευρώπη αυτή η κατάσταση και πώς η Ένωση συνεισφέρει σε αυτό το στόχο του ελέγχου των ε, πυρηνικών. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω και εγώ αγγλικά από, την, από το EUISS. Έχουμε, όπως ξέρετε, τη διάσκεψη για την εξέταση της μη διάδοσης, της συνθήκης της μη Θα προσπαθήσω να καλύψω κάποια ζητήματα που δεν κάλυψαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι και κυρίως ο κύριος Χίψ ε, που εστίασε στα θέματα του Ιράν. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το προφίλ ε, της Ένωσης ως πρωταγωνιστά θέματα ελέγχου όπλων ή μη διάδοσης. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τέσσερις άξονες βασικά. Ένα είναι να συνεισφέρει στην επίλυση κρίσεων για τη διάδοση ποινικών. Δεύτερο, να συντονίσει τις θέσεις και να προσπαθήσει να διατηρήσει ζωή αυτή τη συνθήκη. Επίσης, να προωθήσει οικουμενικές συνθήκες ε, καθολικής ε, ισχύω και να παράσχει οικονομική υποστήριξη σε προγράμματα μη διάδοσης ε, και αποπυρηνικοποίησης. Μια έτσι πρόορια αξιολόγηση του ρόλου της Ένωσης στους δύο βασικούς τομείς δράσης ή e τη συντονισμό για τη συνδική μη διάδοσης και επίλυση κρίσης ε, στον τομέα της διάδοσης είναι ότι τα πάει πιο καλά στο συντονισμό, στο πλαίσιο του NPT, της NPT και όχι τόσο στην αντιμετώπιση κρίσεων. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση δημοσιοποιήθηκε το 2003 που συνέπιπτε χρονικά με τη δρομολόγηση της στρατικής της Ένωσης για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Μέχρι το 2015 είχε συμβεί σχεδόν το αντίθετο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποδειχθεί να είναι αποτελεσματικός παράγων ε, στην επίλυση της κρίσης του Ιράν, για παράδειγμα, που ήταν ε, και μείζον επίτευγμα και στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Όμως, στη διάσκεψη αναθεώρησης του 2015, σε σχέση με την σύμβαση, τη συνθήκη τη μη διάδοση, δεν κατέληξε σε κοινή θέση και εκεί μάλιστα ε, υπέστη και ήττα. Άρα είδαμε να αντιστρέφονται τα πράγματα σε σχέση με την πρώτη, πρώτη αξιολόγηση, την πρώτη αξιολόγηση που είχε γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θεωρείται ότι έχει ένα θετικό ρόλο ε, διότι ακριβώς έτεφα το συντονισμό των κρατών μελών που είναι τόσο διαφορετικά ως προς τις προσεγγίσεις που έχουν ήταν κάτι θετικό. Δηλαδή η Ένωση φαινόταν ότι μπορεί να δημιουργήσει συναντικές θέσεις που θα εξήγαγε έπειτα ε, στο ανομογενές διεθνές πλαίσιο. Μέσα σε μια μικρή ομάδα χωρών της ΕΕ, δηλαδή έχουμε πυρηνικές δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία, αλλά και πολύ ένθερμους υποστηρικτές ε, του αφοπλισμού, όπως είναι η Αυστρία και η Ιρλανδία. Και βέβαια έχουμε και μια μεγάλη ομάδα χωρών που καλύπτονται από την ε, γκέης πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί, με μάλλον παρουσιάζει θέσεις ε, και καταθέτει έγγραφα ε, εργασία ω Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνδίκη μητάσεω. Όμω και μεμονωμένα τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν δηλώσει και να υποβάλουν ε, working papers. Και όλα αυτά δεν αποκλείουν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλου ομίλου. Όπω είναι η πρωτοβουλία για τη μη διάδοση αφοπλισμού, όπω είναι η Πολωνία, η Ολλανδία, η Γερμανία. Ή έχουμε νέου συνασπισμού. Μια τα Έχουμε λοιπόν έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον στερέωμα που είτε μέσω της Ένωσης είτε μέσω άλλων ομάδων μπορούν τα κρατημέλη να ε, δρουν και να αποφασίζουν. Τι έγινε λοιπόν σε επίπεδο συντονισμού στην τελευταία έκδοση της διάσκεψης για την ε, εξέταση της ε, συνθήκης. Από το 1995 είχε τη συνήθεια να καταλύσει κοινέ θέσει η Ένωση, συμφωνώντα σε αριθμού αριθμού προτεραιοτήτων και προπαρασκευάζοντα τη διάσκεψη του 1995... είχε καταλήξει με κοινή θέση ακριβώ η Ένωση, που ουσιαστικά ήταν ένα μονοσέλιδο με πολύ βασικά σημεία. Το ίδιο έγινε στην επόμενη συνεδρίαση ε, εξέτασης που έγινε το 2000. Μέχρι το 2005 τα ουσιαστικά αυτά σημεία συμφωνίας είχα φτάσει τις τέσσερις σελίδες. Η κοινή θέση λοιπόν της Ένωσης πλέον ήταν τετρασέλιδη και το 2010 η κοινή θέση έφτασε στο ρεκόρ των έξι σελίδων κοινών συστάσεων που βλέπουμε ε, να δείχνει εκθετική αύξηση ε, της δυνατότητας συνένεσης ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Τι έγινε όμως το 2015. Το 2015 δεν υπήρξε καν κοινή θέση. Ανταυτού υπήρχε ένα έγραφο με κάποιες προτάσεις και κάποια συμπέρασμα του Συμβουλίου. Ξέρουμε όμως ότι είναι διαφορετική η κοινή θέση που είναι ένα νομικά θεσμευτικό μέσο από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που είναι πολιτικά ε, πιο πολύ. Συνιστούν πολιτική δέσμευση. Και το περιεχόμενο των συμπερασμάτων ήταν πιο έτσι, ασαφές και πιο αδύναμο από ό,τι ήθιστε να βλέπει κανείς ε, στις κοινέ θέσεις του Συμβουλίου. Και βέβαια έρχομαι στο ερώτημα που μας απασχολεί τι, όλους, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τη διαδικασία της ε, συνθήκης με διάδοση να την υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία κτλ βασικός στόχος και σαφής στόχος της Ένωσης είναι ότι θέλει να διατηρήσει εξ ολοκλήρου αυτή τη συνθήκη και αυτό είναι και επιτακτική ανάγκη να γίνει. Γιατί η όλη η διαδικασία ε, είναι βάλωτη αυτή τη στιγμή, είναι σε κρίση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή την ε, πολιτική της ε, υποστήριξης της πολυμερούς προσέγγισης. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει μια στρατηγική που θα καταφέρει να ενισχύσει τη συνθήκη για τη μη διάδοση στην επόμενη διάσκεψη εξέταση. Τι μπορεί να γίνει για το σκόπο αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 2015 κατέστη σαφέ πω η Ένωση δεν είναι πλήρω ενωμένη σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό. Ο εσωτερικό συντονισμός ε, της Ένωσης για την επίτευξη συνένεσης είναι κάτι πρέπει να συνεχιστεί και είναι μια πολύ χρήσιμη άσκηση για την πιέση στα κράτη-μέλη ε, στην αναζήτηση συνένεσης και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί το εγχείρημα αυτό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να είναι πιο επιλεκτική και να κοινέ δηλώσεις να καταθέτει κοινά έγγραφα εκεί που υπάρχει συμφωνία ισχυρή. Και όταν οι προτάσει αυτέ έχουν να προσθέσουν κάτι, έχουν προσθέμενη αξία για την όλη διαδικασία. Αν υπάρχουν τέτοιε ισχυρέ συμφωνίε ή προσθέμενε αξίε, αν δεν υπάρχουν μάλλον αυτά, μπορεί να ακολουθεί μια άλλη προσέγγιση μέσω άλλων ομάδων, όπως το MPDI για παράδειγμα. Ή το New Agenda Coalition. Δεύτερη πτυχή που πρέπει να απασχολεί στην Ένωση αν θέλει να κάνει έτσι μια πιο θετική συμβολή είναι ουσιαστικά πιο πολύ αυτό αποτελεί σύσταση προς τα κράτη-μέλη και όχι τόσο για το Συμβούλιο, αλλά έχει τόσο και για το Συμβούλιο. Προσπαθήσει λοιπόν η Ένωση να βρει ένα μόντους βιβέντη με τη συνήθεια αποκλεισμού. Υπήρξαν ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και αυτή η σχετική αποκλεισμή ήταν η βάση της συμφωνίας. Πώς αυτή η συνθήκη απαγόρευσης αποκλεισμού όταν τεθεί σε ίσχυ. Πώς μπορεί να ε, εννοηθεί, να εννοηθεί ως ανταγωνιστική συνθήκη ή σε πληρωματική συνθήκη προς την συνθήκη με διάδοση των όπλων. ουσιαστικά να παροτρύνει τα κράτη που έχουν υπογράψει την συνθήκη μη διάδοση να, κάνουν, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Η Σουηδία είχε καταθέσει μία πρόταση ένα εφαλτήριο και φαίνεται ότι τα περισσότερα κράτη θέλουν να προχωρήσουν με τον αφοπλισμό. Ενώ τα συμβαλόμενα μέρη της Είπα ότι ε, θα μπορούσαν οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ένωσης να εξαχθούν και σε ένα πιο διεθνές πλαίσιο. Αλλά υπάρχει μια διαφορετικότητα ε, και πολυμορφία. Κυρίως όμως η πλειοψηφία ε, εκεί γέρνει πλάστικα, ενώ στη, στο διεθνές επίπεδο μπορεί να γύρει και προς τη μεριά μιας μειοψηφίας. Το θέμα είναι ποιος είναι ο προσανατολισμός των περισσότερων. Και στις δύο περιπτώσεις δεν συμπίπτουν αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ε, Rebecca Johnson. Ε, του Ινστιτούτου Αφοπλισμού και πρόεδρος της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών. Θα μας παρουσιάσετε την άποψή σας για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό και το δυναμικό αλλά και τα όρια της δράσης της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Είμαι περήφανη Ευρωπαία, έτσι σας μιλάω σήμερα. Η πρώτη φορά που ψήφισα ως το 1975 ως νεαρή φοιτήτρια ήταν για να επιβεβαιώσω ε, την ε, ένταξή μας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά θλίβομαι για αυτό που συμβαίνει. Αυτό μας θυμίζει ότι όταν υπερφύαλοι ηγέτες παίζουν πολιτικά παιχνίδια όταν δεν έχουν σκεφτεί πραγματικά μέχρι τέλους όλες τις ε, συνέπειες, δεν ελέγχουν κατά ανάγκη και αυτές τις συνέπειες. Η Βρετανία που έφυγε από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη. Μην το ξεχνάτε λοιπόν όταν ακούτε και σκέφτεστε τα πυρηνικά, κάτι που κάνουμε σήμερα. Θα ήθελα να μιλήσω για τέσσερα βασικά στοιχεία. Ε, Δυστυχώ οι προλαλήσαντες μίλησαν και αυτοί γι' αυτό. Μπορώ να τα διατρέξω εντάχει. Θέλω να μιλήσω για την NPT, τη Συνθήκη Μη Διάδοση των Πυρηνικών. Ε, ευχαριστώ την Άγγελα που μας είπε πολλά για το που έχουμε φτάσει σήμερα. Έχω φτάσει σε κάθε συνεδρίαση της ε, διάδοσης NPT από το 1994 και την προσπάθεια επέκταση του 1995 και όλες τις προπασκευαστικές συνεδριάσεις ε, και τις διασκέψεις ε, για την αναθεώρηση. Θα ήθελα να σας πω ότι μπήκε, σε ισχύ, τέθηκε σε ισχύ το 1970 με πέντε ε, κράτη που είχαν πυρηνικά 40.000 όπλα, κυρίως οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι τα είχαν. 50 χρόνια μετά ο αριθμό έχει ε, μειωθεί. 13.800 ε, είναι τα πυρηνικά όπλα με βάση το ΣΥΠΡΙ, το Ισουδικό δηλαδή Ινστιτούτο, αλλά τα περισσότερα ανήκουν, ανήκουν πάλι στη Ρωσία και στι ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τώρα εννέα ε, κράτη που έχουν πυρηνικά. Και θα ήθελα να τονίσω ότι μιλάμε για τα βασικά κράτη που επιλέγουν αν θα εκτοξεύσουν ή όχι τα όπλα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό όταν σκεφτόμαστε τον αφοπλισμό, αν το θέλουμε ή όχι. Εννέα ηγέτε στον χώρο των πυρηνικών. παρά το γεγονό ότι έχουν μειωθεί σε αριθμό τα πυρηνικά, το οποίο είναι θετικό. Σε ανθρωπιστικού όρου, ε, ο διπλασιασμό ε, των κρατών που έχουν πυρηνικά αυξάνει τον κίνδυνο. Ε, τον κίνδυνο της χρήση των πυρηνικών, των ατυχημάτων και των πολέμων. Έβαλα εδώ κάποια στοιχεία στην διαφάνεια που νομίζω ότι καλό είναι να μην τα ξεχνάμε. Ε, κοιτάξτε αυτό το θέμα για να δείτε ποιες είναι οι προκλήσεις, για να δείτε ποια ήταν η πορεία, ειδικά από το 1995 και μετά, όταν έγινε μόνιμη η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών, αλλά θα εστιάσω κυρίως σε αυτό το άρθρο, το άρθρο 6 για τον αφοπλισμό, που κοιτάει τρία στοιχεία. Την ανάγκη να σταματήσει η κούρσα των εξοπλισμών, από ό,τι φαίνεται, όμως, επιστρέφουμε σε μιακούς εξοπλισμών μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Δεν έπρεπε δεν, να γίνει, δεν ήταν ανάγκη να γίνει και όμως συμβαίνει. Ακούσαμε πάρα πολλά από την Άγγελα Κέιν για το θέμα αυτό. Ε, και η δέσμευση για την, τον πυρηνικό αφοπλισμό 50 χρόνια είχαν τα κράτη για να το υλοποιήσουν αυτό. Όλα αυτά τα βήματα, όλες αυτές οι όλα αυτά τα λιθαράκια που είχαν μπει, ε, όλο το πλαίσιο για τον πυρηνικό αφοπλισμό που είχε τεθεί, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία, όλες αυτές οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν συζητηθεί ξανά και ξανά, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί από τις βασικές χώρες που έχουν το βασικό ρόλο στην εφαρμογή. Γιατί είναι οι χώρες που έχουν τα πυρηνικά όπλα. Επομένως θα πρέπει να το κοιτάξουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο όπου έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Πούτιν, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι ή να παραβιάσουν τις συνθήκες ε, στις οποίες έχουν ενταχθεί ή να αποσυρθούν από συνθήκες και να καταργήσουν τα νομικά καθεστώτα που μας έδιναν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των πυρηνικών. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν, μέσα στο οποίο ε, κινούμαστε, το ε, παρουσίασε και η Άγγελα, ε, στον προϋπολογισμό του 2021 έχουμε νέα πυρηνικά όπλα στην Αμερική, το είπε ο Τραμπ, ε, ενισχυμένα πυρηνικά και όλα αυτά τα συστήματα ε, είναι πολύ επικίνδυνα, πολύ αποσταθεροποιητικά για την Ευρώπη. Ε, υπερχητική πύραυλη. διαβάσαμε στο New York Times ότι αναπτύχθηκαν ως ανταπόκριση στο πρόβλημα της πυραυλικής άμυνας. Ε, έχουν όμως και απρόβλεπτη πορεία. Ε, έχουμε τέτοια όπλα και έχουμε και μια νέα γενιά ε, πυράβλων κρούς ε, εκτόξευση από το έδαφος που δοκιμάζονται τώρα, τις, ε, κάνει δοκιμές και η Ρωσία και η Αμερική κάνει, επενδύει σε μια νέα γενιά πυράβλων κρούς. Έχουμε λοιπόν όπλα τα οποία μπορούν να μην λειτουργήσουν σωστά και μιλάμε για όπλα μεσαίου ε, βεληνικούς. Ε, τη δεκαετία του 80, όταν ήμουν ακτιβίστρια, που δούλευα για τη συνθήκη για πυρηνικά μεσαίου βεληνικούς, αυτά τα όπλα τώρα έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν στην Ευρώπη θέατρο επιχειρήσεων, θέατρο πολέμου. Οι Αμερικανοί λένε ότι με τη χαμηλή απόδοση αυτών των όπλων, τις νέες πυρηνικές κεφαλές, τις νέ, τη νέα γενιά όπλων, ε, το W87, το πρόγραμμα τροποποίησης, είναι πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να σας κάνουν να σκεφτείτε «Α, μια και δεν έχουμε τώρα 100 κιλοτόνους, αλλά χαμηλό, πιο μικρές ας πούμε, πυρηνικές ε, κεφαλές, έχουμε 5 με 7 ας πούμε, κιλοτόνους ε, σε κάθε πυρηνική τόσο ζυγίζει κάθε πυρηνική κεφαλή. Αλλά με αυτή τη στρατηγική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο εύκολα τα πυρηνικά όπλα. Και θα πρέπει να γνωρίσουμε τελικά ότι η αποτροπή δεν είναι ο σκοπός των πυρηνικών όπλων ή δεν είναι κάτι στο οποίο πιστεύουν οι ηγέτες. Δεν πιστεύουν στην αποτροπή. Και δεν θα πρέπει να πιστέψουμε κι εμείς ότι λειτουργεί αυτή η αποτροπή. Αυτά τα νέα ενισχυμένα λοιπόν, πυρηνικά όπλα από τα κράτη με πυρηνικά δείχνουν ότι δεν δουλεύει η πυρηνική αποτροπή. Επίσης, οι στρατιωτικοί δεν τους αρέσει, δεν, δεν αρέσκονται στην ιδέα της αποτροπής. Και σίγουρα δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά για πολέμους. Αυτά ε, τα ακούμε σε διάφορες ε, στρατιωτικές ακαδημίες, αλλά έχουμε να κάνουμε με μονόθαλμους ηγέτες που δεν μαθαίνουν από την ιστορία και τον ψυχρό πόλεμο. Ε, ότι δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να, δω να δώσουμε τη μάχη με τα πυρηνικά, ότι δεν πρέπει να υπάρξει πυρηνικό πόλεμο. Θα πρέπει, επομένω, να μην αναπτυχθούν στην Ευρώπη ούτε παλιά ούτε νέα συστήματα ε, πυρηνικών όπλων, ούτε υπό το ΝΑΤΟ, ούτε υπό καμία άλλη πλατφόρμα. Ε, έχουμε αυτό το W76, αυτέ τι νέε πυρηνικέ κεφαλέ. Το, το Πεντάγωνο λέει ότι έχει προβλήματα λογισμικού με αυτέ τι πυρηνικέ κεφαλέ. Αυτή είναι κίνδυνη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και μία γρήγορη δράση απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε και τους ανθρωπιστικούς ε, κινδύνους και τους κινδύνους ε, ασφαλείας, ε, γιατί μπορεί την Ευρώπη να την κάνουμε, να την καταστήσουμε μία πυρηνική αμυντική συμμαχία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και οι βουλευτέ θα πρέπει να παίξουν ηγετικό ρόλο για να προωθήσουν ψηφίσματα, αποφάσει και νομοθεσία για να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν την, το καθεστώ μη διάθωση ως βασικό δίκτυο ε, μεταξύ συνδεδεμένων ε, νομικών εργαλείων που θα δημιουργήσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο και θα μας εξασφαλίσουν τον αφοπλισμό. Θα πάω στη συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων. Ε, άρθρο 6 ε, της Συμφωνίας NPT και αυτή η συμφωνία υλοποιεί την... Συγγνώμη, αυτή η συμφωνία ε, εδράζεται στο άρθρο 6 της NPT. η NPT, η συνθήκη για τα χημικά, η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών έτυχαν διαπραγμάτευσης ως στα πλαίσια μιας συνθήκης για ανθρωπιστικούς λόγους, όπου οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις τίθενται στο επίκεντρο και οι ανάγκες των αμάχων επίσης τίθενται στο ε, ε, επίκεντρο. Βασίζονται στο καθεστώς της NPT, αλλά σκοπό έχει να καλυφθούν όλα τα κενά της NPT για, την, για τον αφοπλισμό. Η NPT δεν απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή και την κατοχή πυρηνικών όπλων. Παρότι στο προήμιο τονίζει ότι ο σκοπός της είναι να αποτρέψει τον ε, κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Ε, η συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών και η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών απορρέει από την NPT και απαγορεύει όμως τη χρήση και την απειλή πυρηνικών όπλων, καθώς και όλες οι σχετικές δραστηριότητες αγοράς, ε, παραγωγής, κατοχής, ε, δοκιμών και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, που είναι η προπομπή για πυρηνική αγορά και χρήση. Πυρηνικές αγορές και χρήση. Επομένως, Αυτές είναι οι βασικές απαγορεύσεις που έχει η συνθήκη και καλύπτει και την κατοχή, ανάπτυξη, καθώς και τη βοήθεια. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, η απαγόρευση της βοήθειας, ενθάρρυνσης και προτροπής ε, καθιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε, να προωθήσει δράσεις που απαγορεύονται από τη συνθήκη, αυτό αφορά και μη κρατικού φορείς και εταιρείε. Ε, στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε ότι οι κρατικοί φορεί θα πρέπει να εφαρμόσουν τι υποχρεώσει τη συνθήκη και να σεβαστούν τις, ε, και να σεβαστούν μάλιστα και τη συνθήκη όλα τα άτομα, ε, φορείς και τα λοιπά που είναι υπό τον έλεγχό τους. Υπό τον έλεγχό τους. Η θέση σε ισχύ θα γίνει μάλλον κατά τέλη του 2020 ή αμέσως μετά. Η συνθήκη επίσης απαγορεύει, απαιτεί την πλήρη εξάλληψη και μιλάει για τη διαδικασία εξάλληψης καθώς και τις διαπραγματεύσεις ε, που πρέπει να κάνει μια χώρα που έχει πυρηνικά όπλα που έχει στην επικράτειά της ε, πυρηνικά όπλα. Ε, τονίζει λοιπόν ποια είναι η δημοκρατική διαδικασία για να ενταχθεί στην συνθήκη. Θα ήθελα να πω τα τελευταία μου λόγια στη σημασία για την σημασία των ηθικών, όχι για τον αφοπλισμό, αλλά γιατί είναι γενικά σημαντικές οι συνθήκες. Ε, έχω βεβαίως και άλλες παρατηρήσεις που μπορεί να τις δώσει η γραμματεία, ε, παρατηρήσεις υπέρ των συνθήκων, understand, but I, I, I think I only had, had, had... Ε, τώρα έκλεισα τα 10 λεφτά εδώ. Είχα πολλά ακόμα να πω. Ε, θέλω να πω τι μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτές, τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες για να υποστηρίξουν την NPT, τη συνθήκη μη διάδοσης μέσα στο 2020 και την ε, διάσκεψη αναθεώρησης και την ευρωπαϊκή ασφάλεια ποικιλοτρόπως γιατί έχουμε ανησυχητικέ νέες εξελίξεις για τα πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ. Merci, merci beaucoup pour ces interventions très... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, τόσο πλούσια παρέμβαση. Δεν είμαστε όμως σε πανεπιστήμιο, είμαστε σε κοινοβούλιο και πρέπει να μπορέσουμε να ακούσουμε και τους βουλευτές και το τι έχουν να πούνε και να θέσουν και ερωτήσει ε, και να κάνουν και παρατηρήσεις. Και ο στόχος είναι επίσης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ο διάλογος σε αυτές τις συναντήσεις. Και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μίξερ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες που είναι και εισηγητής ε, για τα θέματα της μη διάδοσης ε, πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω πολλέ ερωτήσει, αλλά θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε κάποιε πολύ συγκεκριμένε, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Καταρχάς, όσον αφορά τη συνενετική θέση των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον πυλώνα της ε, χρήσης πυρηνικών ε, τη Συμφωνίας Μη Διάδοσης, επειδή ήμουν και υπουργό εξωτερικός της χώρας μου για πάνω από δύο χρόνια και σε αυτό το πλαίσιο έχω βρεθεί και στο τραπέζι του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας πω ότι η πολιτική εξωτερικής ασφάλειας είναι και <clears throat> αποκλειστικός ρόλος ε, της ε, διακυβερνητικής συνεργασίας. Εμείς έχουμε βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω από 700 ερετούς οι οποίοι ε, εκπροσωπούν τις χώρες τους και δεν φυσικά απαραίτητο από τις ε, θέσεις ε, στο Συμβούλιο ή τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε δεν είναι δεσμευτικά λόγο αυτό. Είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι εδώ. Όσον αφορά τώρα την πολιτική χρήση πυρηνικών και των πυλών αυτό, uh, υπάρχει μια συζήτηση που αφορά τα θέματα ενέργειας εδώ στο Κοινοβούλιο που εν μέρη έχει και επικαλύψεις με τη συζήτηση για τη μη διάδοση, αλλά κυρίως είναι ξεχωριστή από αυτήν. Είναι μια συζήτηση για τα περιβαλλοντικά και για το κλίμα που είναι ε, μια από τις ε, βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αυτού για αυτή τη θητεία. Ορισμένες φορές αυτές οι συζητήσεις ε, ε τείνουν να σκιά, επισκιάζουν την ε, ε, αναθεώρηση της συμφωνίας με διάδοση και τη σχετική διάσκεψη. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα περισσότερα πράγματα όσον αφορά το πώς ο πυλώνας ε, ε πολιτικής χρήσης ε, της, ε, των πυρηνικών έχει κάποιε διαστάσει. Παρά το γεγονό ότι δεν είναι ρηπογόνο ε, η πυρηνική ενέργεια προ τον άνθρακα, τείνουμε να την ε, δαιμονοποιούμε γιατί δεν θεωρείται ότι είναι περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο παραγωγή ενέργεια. Αλλά στα πλαίσια όμω τη ε, ε συμφωνία μη διάδοση, κυρίω εξετάζουμε την μη διάδοση και όχι την περιβαλλοντική πτυχή τη ενέργεια και την παραγωγή πυρηνική ενέργεια. Μια δεύτερη ερώτηση, σχόλιο για τις προσπάθειες να στιγματίσουμε όλα τα πυρηνικά όπλα. Φοβάμαι ότι ακόμα και αν ε, η συνθήκη έχει αυτό το στόχο και δεν ε, συλλάβουν νόμιμα με ε, τα όσα αποφασίζονται, εγώ θα προτιμούσα να μην δημιουργήσουμε μία ψευδή ισότητα μεταξύ των πέντε πυρηνικών κρατών και ε, των ανθρώπων που είναι εκτός της συμφωνίας, δηλαδή το τι πρέπει να κάνει η Βόρεια Κορέα ή το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ έχει και μία συμμαχία για τα πυρηνικά και λέει ότι είναι ε, υπέρ ενός ε, ε, κόσμου χωρίς πυρηνικά, αλλά όσο υπάρχουν πυρηνικά θα παραμένει και πυρηνική δύναμη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια δημοκρατική, υπεύθυνα η ε, πολιτική για τα πυρηνικά για να κλείσουμε το διακόπτη για τα πυρηνικά όταν θα φτάσουμε σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επιστρέψω και σε κάτι που είπε και η κυρία Κέιν όσον αφορά την ευρεία υποστήριξη. Εμένα δεν με εκπλήσει το 80% της στήριξη των νέων, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρω ότι κάποια μη δημοκρατικά κράτη είναι πάρα πολύ περήφανοι για τις πυρηνικές τους δυνατότητες σε επίπεδο κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι και οι πολίτες τους ε, είναι και λιγότερο αντίθετοι στις πυρηνικές κανότητες της χώρας. Πώς μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ της ε, άποψης ε, της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης και της ρωσικής κοινή γνώμης. Ευχαριστώ, Μαϊκ για την ΚΟΕ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον καθένα από εσά να μιλάει για 1,5 λεπτό, γιατί αλλιώ δεν θα έχουμε χρόνο για τι απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Κάποιες σύντομες ερωτήσεις κυρίως προς την Άντζελα και τον κύριο Χίπς, ε, του οποίου μου διαφεύγει το μικρό του όνομα. Αναφερθήκατε στη ε, κλιμάκωση στις δαπάνες. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι δαπανάουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι οι Ρώσοι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση των δύο. Δεύτερον, η πίεση να αυξηθεί η δαπάνη από πού προέρχεται πιο συγκεκριμένα κατά την άποψή σας. Πολύ συχνά Βλέπουμε προσπάθειες ε, να αυξηθεί η πυρηνικοποίηση στην Ευρώπη έχει και σχέση με τη ε, αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Από πού προέρχονται λοιπόν οι πιέσεις. Τρίτον, Νομίζω το πιο τρομακτικό που έχουμε δει είναι η νέα βόμβα που είναι αρκετά μικρή για να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας θεωρείτε ότι και άλλες χώρες πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν ε, και να επεκταθούν στον τομέα αυτό. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να διαδοθεί συγκεκριμένη βόμβα. Τώρα, η συμφωνία με το Ιράν. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα μέλο, οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν από τη συμφωνία και δεν θέλουν να ξέρουν τι γίνεται. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να συνεχίσει, ε, υπάρχει θετική στάση από πλευρά Ευρωπαίων, είναι αβοήθητοι, μπορούν να κάνουν περισσότερα χωρί τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μια τελευταία ερώτηση. Όταν ε, συζητούμε για πυρηνικές απειλές και μη διάδοση όπλων ε, και λοιπά και κανόνες και ένα κόσμο βάσει κανόνων, αυτό που δεν αναφέρεται είναι το Ισραήλ. Πώς βλέπετε τη δική τους τη θέση σε όλο αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Γκροσίλη από την ομάδα Renew Europe. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω απλά είναι τα πράγματα δύο θέσεις υπάρχουν στον κόσμο. Ότι η συνθήκη για τη μητέρα των όπλων είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί, αλλά η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Έχουμε την INF για τα όπλα μικρού βελληνικού. έχουμε μέσου έχουμε τη συμφωνία για το Ιράν που καταργούνται. Άρα εύκολη κατάρρευση μια συμφωνίας, δύσκολη δημιουργία νέα ε, συμφωνία ή συνθήκη. Εγώ κάπως κατανότηση είπα, γιατί ξέρω τι φοβούνται ε, με τις συζητήσεις ε, για την ε, σύμβαση. Αν γίνει πυρηνική δύναμη το Ιράν, ακολουθεί Σαουδική Αραβία κτλ. κτλ. Τα Ενόμενα Αραβικά Εμμυράτα και ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες όπως το Πακιστάν που εξάγει πυρηνική τεχνολογία, που ήδη έχουν πυρηνικά όπλα. Για την Ευρώπη και για τη Δύση βέβαια εν γέννη. Το θέμα είναι πώς από τη μία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αποτροπή και από την άλλη να ξεκινήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κάτι ανάλογο με τη δεκαετία του 80, όταν είχαμε αυτή τη συμφωνία του ΕΝΕΦ για τα πυρικά όπλα μέσω βελληνικούς και τη συμφωνία περί αφοπλισμού. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αρκέσει η αποτροπή και το βλέπουμε ήδη αυτό. Αν η άλλη πλευρά βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, θα έχουμε ξανά κούρσα πυρηνικών όπλων. Ρωσία, Κίνα, ΙΠΑ, σε κάποιο βαθμό έχουν ήδη μπει σε αυτή την κούρσα. Ε, έχουμε τις νέες τεχνολογίες, ε, υπηρχετικούς πυράβλους, ε, αυτές τις βόμβες χαμηλής απόδοσης στις τρεις χώρες αυτές. Η χρήση λοιπόν πυρηνικών όπλων, το κατόφλι έχει χαμηλώσει πολύ. Έχουμε 9 κιλοτόνους ε, και τρομερή αύξηση της τεχνολογίας. Το ποσοστό σφάλματος πριν 10-20 χρόνια υπολογίζονταν σε χιλιόμετρα ε, οι δεκάδες χιλιόμετρα και τώρα σε μέτρα, οι δεκάδες μέτρα. Και Ιράν και άλλες χώρες έχουν τη δική τους λογική. Θεωρούν ότι αν έχουν πυρηνικά όπλα θα είναι ασφαλείς. Άρα αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Πώς θα τους πείσουμε ότι θα είναι πιο ασφαλείς χωρίς πυρηνικά. Και απ' την άλλη πώς θα αποτρέψουν τις χώρες αυτές, ώστε να μην συνεχίσουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Merci pour les για τους Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες Πραγματικά μας ε, δώσατε πολύτιμη ε, γνώση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ε, άκουσα κάπως με ανοιχτό στόμα κάποια επιχείρηματα για τη στρατιωτική και μη στρατιωτική χρήση των πυρηνικών. Εγώ πιστεύω ότι ο φόβος της πυρηνικής ενέργειας για το ενεργειακό μείγμα ε, δεν είναι και τόσο μεγάλος. Δεν θα φτάσουμε στην ανάπτυξη ενός μη πυρηνικού όπλου γιατί είναι, για να σώσουμε το κλίμα άμεσα. Ξέρουμε πόσα χρόνια χρειάζεται έρευνα. Στη Γαλλία έχει αποτύχει και οι λομπίστες που προωθούν ε, την πυρηνική ενέργεια ουσιαστικά θέλουν να βάλουν και τη σφραγίδα του πράσινου συμφώνου για να συνεχίσουν να ε, έχουν τα κέρδη και να ευημερούν. Όποιοι μπορούν θα θα δημιουργήσουν ε, στρατιωτικά ε, πυρηνικά όπλα μέσα από τον ε, μη στρατιωτικό τομέα. Υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχει η Ινδία, χώρες που έχουν έτσι ξεκινήσει και έτσι έφτασαν στα πυρηνικά όπλα. Θα ήθελα να μου πείτε για τον τρίτο πυλόν. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμος και αν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε να έχουμε αυτό το μη στρατιωτικό όπλο και να το επιτρέπουμε σε κάποιες χώρες, δεν οδηγεί αυτό κάποια στιγμή και στη μοίρα στρατιωτικών όπλων. Για το κατά πόσον είναι συμβατές οι δύο συνθήκες ή όχι. Για, τον, για την απαγόρευση ή για τη μη διάδοση. Εγώ έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Ναι, όμως ισχύει πράγματι και αν ναι σε ποιο άρθρο εδράζεται. Και το διεθνές δίκαιο, παρά τους δεν είναι η λύση για να βγούμε από το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τη μη διάδοση. Θα ήθελα να έχω μια νομική απάντηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασέσκου τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια παρατήρηση και μετά μια ερώτηση. Η παρατήρηση αφορά τη μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Και για να είμαι ειλικρινή, αν θέλουμε να έχουμε μια επιτυχημένη πράσινη συμφωνία, δεν θα το πετύχουμε χωρίς πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα και τους υδρογονάνθρακες και την πυρηνική ενέργεια να τα καταργήσουμε ταυτόχρονα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική χρήση. Νομίζω ότι ε, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ανεχόμεθα το Ιράν. Και το κάναμε ακόμη και όταν το γνωρίζαμε και μας το είχαν ήδη πει ότι οι Ιρανοί δεν καταθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να πείθουν ότι δεν συνεχίζουν το στρατιωτικό τους πρόγραμμα. Από αυτές ε, τις συνθήκες, νομίζω ότι τα δημοκρατικά κράτη δεν έχουν δικαίωμα να επιτρέπουν σε μια χώρα όπως είναι το Ιράν να αναπτύσσει στρατιωτικά όπλα με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Είναι και το σφάλμα που έγινε με τη Βόρεια Κορέα. Το ίδιο λάθος έγινε. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Αν το Ιράν δεν σεβαστεί τις δεσμεύσεις του, και νομίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν δίκιο, το πιστεύω αυτό, πώς μπορεί να σταματήσει το πρόγραμμα στο Ιράν η κοινότητα. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε το πρόγραμμα. Με διασκέψεις δεν νομίζω. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Αν συμφωνείτε, δυστυχώς δεν έχουμε πλέον χρόνο. Έχουμε 10 λεπτά για να ακούσουμε τις απαντήσεις ε, των ομιλητών μας. Ερωτήσεις για το Ιράν ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορούν συγκεκριμένα το, Ιράκ, το Ιράν και να μπορέσουμε εδώ να επικεντρωθούμε στις ερωτήσεις που ετέθησαν Όσον αφορά την πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, υπάρχουν φυσικά διστάμενες απόψεις μεταξύ των ομιλητών. Ερωτήσεις για τη θέση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τι γίνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν ερωτήσεις όσον αφορά τις δαπάνες πυρηνικά ζητήματα ε, και διαχωρισμός ε, μεταξύ ε, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και τα μικρά πυρηνικά όπλα τα οποία προωθούν. Να κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν και φυσικά υπήρχε και μια ερώτηση για τη συμβατότητα μεταξύ της συνθήκη για την πλήρη κατάρκεση των πυρηνικών όπλων και τη μη διάδοση. Έχουμε 10 λεπτάκια. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ουσιαστικό να επικεντρωθούμε σε αυτά. Να δώσω καταρχά το λόγο στην Άγγελα Κέιν γιατί τι απίφθηνα τι περισσότερε ερωτήσει. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πολύ σύντομα, όσον αφορά τον πυλώνα της, πυρι... της πολιτικής χρήσης. Να υπενθυμίσω ότι είναι ένας πυλώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πάρα πολύ σημαντικός. Δεν αφορά μόνο την ε, πολιτική παραγωγή ενέργειας, αλλά ισότοπα, ιατρικά ζητήματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα λοιπόν που επισέρχονται. Και υπάρχει και μια πτυχή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Ο πρόεδρος Ομπάμα ε, είχε την ιδέα να γίνει μια ε, σύνοδος ε, πυρηνικής ασφάλειας για να μπορέσει να ε, δει και πόσο σημαντικά είναι τα πυρηνικά υλικά υπήρχε ε, πρόσβηξη με πολύ εμπλωτισμένο ουράνιο και χαμηλή εμπλωτισμού ουράνιο. Υπήρχε για παράδειγμα μια πρόταση από το Καζακστάν για να υπάρχει αποθητήριο ε, χαμηλού εμπλωτισμένου ουρανίου για να μπορούν τα κράτη να ζητούν ε, να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για πυρηνική ενέργεια και για ισότοπα κλπ. κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δυστυχώς, το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πυρηνικό υλικό είναι μόνο το 15% όλου του υλικού. Αυτά που είναι λοιπόν σε χέρια πολιτών και όχι για στρατιωτικές χρήσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε και θα έπρεπε. Επίση πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, να σκεφτούμε λοιπόν την πυρηνική ενέργεια γέννη. Αυτό το οποίο συμβαίνει και είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί από εσά ανέφεραν τη Μέση Ανατολή. Όταν σκέφτεστε και άλλε χώρε οι οποίε κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα ή πυρηνικά υλικά. Μία από τι ε, ε περιπτώσει που είναι ψηλά στον κατάλογο είναι η Σαουδική Αραβία δεν θέλουν ε, ε, ουράνιο χαμηλού εμπλωτισμού, θέλουν να κάνουν εμπλωτισμό ουρανίου οι ίδιοι και το δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κατά των διεθνών συμφωνιών, όχι συνθήκη, αλλά διεθνών συμφωνιών. Αλλά δυστυχώ το υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Και υπάρχουν και κάποιε χώρε, και νομίζω ότι οι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα είναι κατά, ε, που θέλουν να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία να ξεκινήσει τη δική της διαδικασία ε, εμπλουτισμού ουρανίου. Όχι να παίρνουν εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά να το έχουν. Έχουν και δεν ξέρω πόσα πυρηνικά εργοστάσια στο Ιράν. Ε, σκέφτονται μπροστά. Όσον αφορά τι υπόλοιπε χώρε στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δεν έχει παραδοχτεί ποτέ ότι έχει πυρηνικά όπλα, αλλά είναι ευρέω γνωστό ότι υπάρχουν. Ε, Ακούγεται κάτι για 30, αλλά είναι ε, δεν είναι σαφές πόσα έχουμε. Το θέμα είναι ότι αν υπάρξουν πιέσεις για τις τέσσερις χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα, τις οποίες γνωρίζουμε, η Βία, Πακιστάν, ε, Ισραήλ και λαϊκή δημοκρατία του Κογκό θα συμμετέχουν ω πυρηνικά κράτη ή όχι. Γιατί η ιδέα είναι ότι συμμετέχει στη συμφωνία ω μη πυρηνικό κράτο. Αυτό λοιπόν δεν έχει προχωρήσει ποτέ και δεν ξέρουμε πώ θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ο πρόεδρο ε, Τραμπ διαπραγματεύεται ε, τη λαϊκή δημοκρατία του Κογκού ω μη πυρηνικό όπλο. Ε, της Κορέα, συγγνώμη. Ε, επομένως, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. δεν έχω τα στοιχεία, δεν μπορούσα να κάνω την έρευνα, αλλά η Σύπρη έχει τα στοιχεία. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά από όσα γνωρίζουμε, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε, γιατί οι πληρώσει που έχουμε από τη Βόρεια Κορέα δεν είναι όσο πλήρη ε, θα θέλαμε. Ε, ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο ε, συντομία να απαντήσει στι ερωτήσει, παρακαλώ. ερώτηση του κ για τον τρίτο πυλώνα. Μην ξεχνάμε ότι οι διαμάχες για τον τρίτο πυλώνα αφορούν τις διαφορές κυρίως μεταξύ των χωρών που πιστεύουν στην προώθηση α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή έχει όρεξη να προωθήσει αυτό το θέμα ε, και στις υπόλοιπες. Το θέμα είναι τι μας ενώνει σε κανονιστικό πλαίσιο. Ε, η μη διάδοση των πυρηνικών είναι ένα στοιχείο ε, που πρέπει να ρυθμιστεί και το άλλο αυτό που είπε η Άντζελα, ε, που είναι η πυρηνική ασφάλεια. Αυτά είναι θέματα που κατά πάσα πιθανότητα ενώνουν τις περισσότερες, αν όχι όλες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ε, κατανοούν την αξία του να έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Είτε μια χώρα είναι υπέρ της πυρηνικής ισχύω, είτε όχι. Αν ε, διαχωρίσουμε το θέμα της ε, προώθησης, ας πούμε, το άλλο που προκύπτει είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ενότητα σε αυτό το θέμα από ό,τι συνειδητοποιεί ο κόσμο. Η Άντζελα μίλησε για τη Σαουδική Αραβία και το μέλλον της. Εδώ τίθεται ένα θέμα που έθεσε και ένας άλλος ευρωβουλευτής. Της, ε, το μέλλον της ε, ειρηνικής χρήσης ε, και τη σχέση ανάμεσα στην ειρηνική και μη ειρηνική χρήση και κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει κατάχρηση της ειρηνικής χρήσης των πυρηνικών. τα, αυτό που μάθαμε από το Ιράν τα τελευταία 20 χρόνια είναι η συνθήκη μη διάδοση δεν εντοπίζει τις, ποιες είναι οι τεχνολογίες για την ειρηνική χρήση. Τι τεχνολογίες υπάρχουν εκεί. Στην περίπτωση του Ιράν και σε άλλες ε, περιπτώσεις άλλων χωρών, ε, ο κύκλος των πυρηνικών ε, καυσίμων και το εμπλουτισμένου ουρανίου ε, σε αυτές τις συζητήσεις που είχαμε για το Ιράν, το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και ο κύκλος του πυρηνικού υλικού ήταν ε, στο κέντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνεισφέρει στη διάσκεψη για την αθεώρηση ε, ότι στα πλαίσια της NPT θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι ειρηνική χρήση. Θα πρέπει να το συζητήσουμε πιο πολύ τα μέλη της συνθήκης αυτό το θέμα για να εντοπίσουμε τις τεχνολογίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, και που θεωρούμε ότι είναι η ειρηνική χρήση. Αυτές είναι οι τεχνολογίες, αυτή είναι η χρήση και θα πρέπει αυτό να το προσδιορίσουν τα μέλη της συνθήκης. Πράγματα τα οποία τι δικαιολογείται και τι όχι. Τα μέλη της συνθήκης, της συνθήκης δεν έχουν κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της μοναδικής της φύσης και του γεγονότος ότι γνωρίζει αυτές τις τεχνολογίες ε, και κατέχει αυτές τις τεχνολογίες, μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία. Ακούστηκαν και άλλες ερωτήσεις με την ειρηνική χρήση των πυρηνικών. Δεν θέλω να τις απαντήσω, αλλά με δύο λόγια να πω το εξής. Η συμφωνία για τα πυρηνικά με το, με το Ιράν ε, μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αβοήθητη, απλώς πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Η εμπειρία της είναι ότι οι οικονομικοί φορείς και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται τις κυρώσεις των ΗΠΑ για το θέμα του, της συμφωνίας με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση για αυτό το θέμα. Τώρα για το μέλλον της συμφωνίας, η συμφωνία λειτουργήσε για πέντε χρόνια. Το Ιράν επί πέντε χρόνια δεν προχώρησε. Το πρόβλημα είναι στο εγγύς μέλλον. Τι θα γίνει. Όταν θα αρχίσει να μειώνεται η ισχύ τη συμφωνίας, να δει η συμφωνία εντό αγωγικών, θα συνεχίζει το Ιράν να σέβεται, η πρόεδρο διακόπτη, δεν έχουμε χρόνο, ε, και σας ε, πρότεινα να μην μιλήσετε, σας είχα πει να μην μιλήσετε για αυτή τη συμφωνία άλλο. Σας δίνω το λόγο για λίγα λεπτά. Ζητώ συγγνώμη που σας ε, κόβω, αλλά αλλιώς θα καθυστερήσουμε πολύ για το επόμενο σημείο. Για τις συνθήκες ε, μη διάδοσης. Διαβάστε όλες αυτές τις συνθήκες και τη συνθήκη της, απαγόρευση απαγόρευσης για να δείτε πού υπάρχουν ασυμβατότητες. Μισή ώρα χρειάζεται για να διαβάσετε και τα δύο έγγραφα. Οι, οι ε, είπαν ότι αναπτύχθηκε αυτή η δεύτερη συμφωνία για να προωθηθεί η συμφωνία για τη μη διάδοση, για το κόστος. Έχω τις λεπτομέρειες ε, από το New York Times για το Trump. Έχουμε 23% αύξηση στον προϋπολογισμό ε, για μη πυρηνικά όπλα σε αντιδιαστολή με την ε, συντήρηση των, ε, των σημερινών όπλων. Αυτά, αυτά μιλάω, αφορούν δηλαδή τους υπηρεχητικούς τα κτλ. Άρθρο 6 της συνθήκης NPT τώρα. Επιπτώσεις ανθρωπιστικές από τη χρήση των πυρηνικών. Αυτό ήταν κάτι που είχε αναγνωριστεί το 2010 τα πλαίσια μια συνένεση στην ε, διάσκεψη της αναθεώρησης. Και η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών τη διαπραγματεύτηκαν 122 ε, χώρες και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιρλανδία, Σουηδία, Αυστρία κτλ. που δεν έχουν πυρηνικά. Ε, σε 122 χώρες είναι και χώρες που έχουν πυρηνικά. Αν είχα περισσότερο χρόνο θα σας μιλούσα για αυτό το καθεστώς, ε, για το πώς αναπτύχθηκε από το 1968 μέχρι σήμερα. Ε, με διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η συνθήκη του 17 του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών είναι μια προσθήκη, πολύ σημαντική στο καθεστώς της συνθήκης μη διάδοσης. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, ε, μας είπε δυο λόγια ο κύριος Σατούρη. Έχετε ίσως δίκιο σε αυτό που είπατε. Προέκυψε από τα δεδομένα για την κατάσταση της ε, πυρηνικής ε, ενέργειας. Μία έκθεση που βγαίνει ετησίως από το Παρίσι και προκύπτει ότι η Κίνα θέλει να προχωρήσει στην παραγωγή, επιπλέον παραγωγή πυρηνικής ενέργειας με τις ε, τεχνολογίες που έχουμε σήμερα, ε, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να σώσουμε και το κλίμα. μπορούμε να κρατήσουμε το, την πυρηνική συνιστόσα στο ενεργειακό μείγμα που έχουμε σήμερα για να διατηρήσουμε το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε την ε, πυρηνική συνιστόσα. Το άρθρο 4 του NPT χρησιμοποιήθηκε ως μηχανισμός ε, διάδοσης τελικά πυρηνικών από πολλές χώρες. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Επίσης, ε, η ελεύθερη ζώνη από πυρηνικά στη Μέση Ανατολή είναι ένα από αυτά τα δύσκολα σημεία όταν ε, συναντηθούν στη Νέα Υόρκη τα κράτη, τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή της συνθήκης για τη μη διάδοση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε για την ε, σύσταση ε, μεταλλόγου Ε, είναι αδύνατο να μιλήσουμε για τη μη διάδοση. Ε, αν δεν μιλήσουμε όλοι ε, και βλέπουμε ότι στο Κοινοβούλιο ειδικά δεν υπάρχει πάνελ εμπειρογνωμόνων χωρίς γυναίκες. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα αργότερα.